πρώτος αντιπρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Δημοκρατίας του Ιράκ. Με χαρά μου θα ήθελα να πω ότι η πρόοδος σε θέματα ασφάλειας και ε, νόμου στο Ιράκ ε, η οποία αποδείχθηκε με τις πρόσφατες εκλογές του Ιανουαρίου είναι τόσο ενθαρρυντικές, είναι πολύ ενθαρρυντικές αυτές, αυτές οι πρόοδοι και ελπίζουμε ότι το Ιράκ πολύ σύντομα θα ξεπεράσει τα δύσκολα χρόνια τα οποία έχει ζήσει τελευταία. Να είστε σίγουροι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό το Κοινοβούλιο θα είναι πάντοτε στο πλευρό σας για να σας βοηθήσουν να ε, εξασφαλίσετε την ειρήνη, τη δημοκρατία και την ασφάλεια. Όλες οι χώρες στον κόσμο και το Ιράκ έχουν δικαίωμα να χαίρουν αυτόν. Ελπίζουμε ότι η επίσκεψή σας θα είναι καρποφόρα και ότι η παρουσία σας θα μας ε, βοηθήσει να εντείνουμε ακόμα περισσότερο τις, ε, τους δεσμούς ε, που μας συνδέουν. Περνάμε την ε, εξέταση σε δεύτερη ανάγνωση, ειδική πλειοψηφία δηλαδή, της κοινής, προ... της του Συμβουλίου για την πρόσβαση στη διεθνή αγορά λεωφορείων και πούλμαν.